προφορική ερώτηση σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επιτρέψτε μου ε, καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας θα πρότεινα να καθυστερήσουμε ένα-δύο λεπτά την έναρξη της συνεδρίασης, γιατί πρόκειται για μια ε, προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχα την ελπίδα ότι ο κύριος Μακρύβη θα είναι παρόν. Α, με συγχωρείτε, είδεν, ε, ε, είναι εδώ ο κύριος Μίχη. Δεν τον είχα ξαναδεί. Είναι εδώ για να απαντήσει εκ μέρους του κύριου Μακρύβη. Εντάξει λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαμέκη. Ε, ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μακρύβη. Ε, πρώτα απ' όλα λοιπόν μεταβιβάστε του τις ε, ευχαριστίες μου. Επίσης ε, χαίρομαι που είναι παρόν ο κύριος Μπάνιε, πολύ ε, ενεργό μέρος της Επιτροπής μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ. Ε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εγκριθεί η, ο διορισμός του από το Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεται εδώ ούτως ή άλλως. Το θέμα το, της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών και της οδηγίας της, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι ένα θέμα για το οποίο ενδιαφέρεται περισσότερο από όλα η Επιτροπή μου στα πλαίσια της οικοδόμησης ενιαίας αγοράς. Και απευθυνόμαστε στην Κομισιόν σήμερα για να ζητήσουμε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο μεταφοράς της ε, ε, αναθεωρημένης ε, οδηγίας ε, του 2005. Πώς εφαρμόστηκε από τα κράτη-μέλη. Και επίσης είναι πολύ επίκαιρη η ερώτηση γιατί ο καθηγητής Μόνση τη Δευτέρα ήρθε στην Επιτροπή μας για να μας μιλήσει για την δική του αποστολή για λογαριασμό του Προέδρου της Κομισιόν σχετικά με τις μελλοντικέ κατευθύνσεις της εσωτερικής αγοράς. Και μας τόνισε ότι ένα μέρος ε, του προβλήματος σχετικά με την εσωτερική αγορά δεν είναι ουσιαστικά η έλλειψη ε, νομοθεσίας. Είναι η συνεπής ε, εφαρμογή των ε, υπαρχών των νομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μα για τη δημιουργία τη ε, ε, εσωτερική αγορά. Για το θέμα τώρα τη αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, όπω πολύ σωστά λέει, πολύ σωστά λέει η διερώτησή μα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ήδη σημαντικά προβλήματα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα προβλήματα θα αντιμετωπίζουν οι πολίτε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει ο μεγαλύτερο αριθμό παραπώνων στα πλαίσια του μηχανισμού Solvit και ε, σε επίπεδο κρατών μελών. Πάρα πολλοί αισθάνονται απογοητευμένοι από την απουσία σαφών ε, αποφάσεων και επίσης λόγω της έλλειψης επαφής ε, μεταξύ των διαφόρων αρχών έγκρισης των διαφόρων κρατών μελών. Η έρευνα που έχει γίνει αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει υπάρχει αρκετή συντονισμένη δραστηριότητα για να βοηθηθεί ε, το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Μία άλλη πτυχή είναι η εξή και είναι επίσης αυτής από τις εργασίες της δικές μας και άλλων, ότι δεν υπάρχουν αρκετά ε, ε αρκετοί επαγγελματίες που σκέφτονται το θέμα αυτό της αναγνώρισης των ε, προσόντους μέσα σε έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν πρακτικά να σκεφτούμε πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό ο μηχανισμό. Και ξέρουμε από τα θετικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή, και σίγουρα θα ακούσουμε τα σχετικά και από την Κομισιόν, ότι η μεταφορά του νομικού αυτού μέσου έχει καθυστερήσει σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, βλέπουμε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι αναμενόταν για να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή. Και σίγουρα αυτό δημιουργεί ανησυχίε σχετικά με την πολυπλοκότητα του νομικού μέσου. Τώρα, για να τα θέσω όλα αυτά στα πλαίσια της ε, ε, εργασία τη Επιτροπή Εθνική Αγορά τα επόμενα πέντε χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ δε που βρίσκονται εδώ όλοι οι συντονιστέ τη Επιτροπή και του ευχαριστώ για τη συνεργασία του ε, για τη διαμόρφωση τη ατζέντα για αυτή την Επιτροπή. Αυτό το θέμα τη ε, αμοιβέ αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είναι ένα θέμα που λύνεται με μια φορά. Ρόλο τη Επιτροπή μα είναι να συνεχίσουμε να ερευνούμε, να προωθούμε και να κάνουμε συστάσει ε, σχετικά με, την, ε, με τις μελλοντικές εξελίξεις των βασικών νομοθετικών μέσων που έχουμε στον τομέα αυτό. Ξέρουμε ότι η Κομισιό πρόκειται να αναθεωρήσει το 2011, να επανεξετάσει την οδηγία αυτή για την αμοιβή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Σχεδιάζουμε συναντήσεις με τους εθνικούς ε, βουλευτές και κοινοβούλια για να συζητηθεί αυτό το πρόβλημα. Θα κάνουμε μια ακρόαση για την υποστήριξη της ε, έκθεσής μας, της αναφοράς μας. Αυτά είναι τα μέσα που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και κάποια στιγμή το 2010 θα συντάξουμε και μια έκθεση πρωτοβουλίας για να τροφοδοτήσουμε τη συζήτηση που θα γίνεται στα πλαίσια της Κομισιόν. Αυτά είναι τα συμφραζόμενα του θέματος αυτού. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τις απάντησεις της Κομισιόν. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας και είμαι σίγουρος ότι ο νέος Επίτροπος θα προωθήσει αυτό το θέμα και θα συνεργαστεί μαζί μας για να προωθηθεί αυτό το κρίσιμο χρήσιμο νομοθετικό ε, μέσο και να βελτιωθεί η εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Επίτροπο Σαμέσκι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για το σημαντικό αυτό ερώτημα και αρχικά θα θέλω να σας παρουσιάσω μία επισκόπηση. Ο στόχος της ε, οδηγίας αυτής αποβλέπει στην ελεύθερη, καλύτερη ελεύθερη διακίνηση ε, των επαγγελματιών στην εσωτερική αγορά. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε δυο κράτη-μέλη και άλλα δύο κράτη ελπίζουμε ότι θα έχουν ε, προχωρήσει. Από την Ελλάδα όμως δεν έχουμε λάβει ακόμη κανένα μέτρο εφαρμογής. Επανέρχομαι τώρα στο πρώτο θέμα. Πρόκειται για μία πρόκληση για τα κράτη-μέλη γιατί εμπλέκει περίπου 800 επαγγέλματα τα επαγγέλματα αυτά μπορεί να έχουν ρυθμιστεί και μέσω ομοσπονδιακών ή τοπικών νομοθεσιών αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για καθυστέρηση και στις ε, έξι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει γίνει αποδεκτή αυτή η προσπάθεια. Ε, ε, τα βασικά προβλήματα λοιπόν αναφέρονται στα επαγγέλματα υγείας και στους αρχιτέκτοντες όπου χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικέ ρυθμίσεις. Επίσης υπάρχουν προβλήματα σε άτομα με, ειδική, ε, ειδικές δεξιότητες όπως η ξεναγή και οι δάσκαλοι. Προσπαθούμε να υπάρξει μία σωστή εφαρμογή της οδηγίας και γι' αυτό έχουμε διαμορφώσει έναν κώδικα συμπεριφοράς που απευθύνεται στους πολίτες για να υπάρχει μια πιο συνεκτική εφαρμογή. Όσον αφορά τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί γνωρίζομαι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ή την διαδικασία αναγνωρίσεως στην εμπλοκή των υπευθύνων αρχών ε, αποφάσεις οι οποίες δεν είναι αιτιολογημένες και ούτω καθεξής και μια φορά δίνεται ακόμη στους μετανάστες λανθασμένη πληροφόρηση και υπόκεινται σε λανθασμένες διαδικασίες. Προσπαθούμε μέσω του Solvit να λύσουμε πολλά από αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν υπάρχει μόνο το Solvit, υπάρχουν τώρα και εθνικά σημεία επαφή σε όλα τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να βοηθηθούν όλοι οι πολίτες και η Επιτροπή θα είναι ακόμη πιο δραστήρια στο μέλλον. Επίσης, ε, ε, το σύστημα εσωτερικής αγοράς έχει καταφέρει να στηρίξει πάνω από 1.200 ανταλλαγές πληροφοριών για ρυθμισμένα επαγγέλματα εφέτος, για βελτίωση της ε, καθημερινής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών. Τέλος λοιπόν, όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει που υπάρχει ανάγκη για προσαρμογή αυτή τη στιγμή. Αυτό θα γίνει σε μία άσκηση εκ των υστέρων που προβλέπεται από την οδηγία. Ε, η Επιτροπή θέλει να γίνει σεβαστή να γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η οδηγία για να δούμε τι μέλη γενέστε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαμέτσκι. Τώρα θα ακούσουμε τις διάφορες παρεμβάσεις για τις πολιτικές ομάδες και καταρχήν για δύο λεφτά θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουρτ Λέχνερ. Ε, ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το 2005 μετά από πολυετή ε, συζήτηση στο Κοινοβούλιο είχαμε ε, αποφασίσει αυτή την οδηγία και εφαρμόστηκε. Τώρα είμαστε το 2009, έπρεπε να ισχύσει από το 2007 και είναι απαράδεκτο η οδηγία αυτή να μην έχει εφαρμοστεί διότι δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, θα ρίνω λοιπόν την Επιτροπή να πιέσει τα κράτη-μέλη είχα φανταστεί ότι θα είχαμε περισσότερα προβλήματα στην πρακτική και αυτό είναι και το αντικείμενο της μελλοντική έρευνας να δούμε δηλαδή πού υπάρχουν προβλήματα επιτόπου και τι συμβαίνει συγκεκριμένα διότι 20% των προβλημάτων στο Solvit αναφέρονται σε αυτό το θέμα και πολύ σωστά είπε ο κύριος Επίτροπος πόσο βασικό είναι το θέμα αυτό για την εσωτερική αγορά από την οικονομική σκοπιά. Είναι ένα ουσιώδες δικαίωμα των ε, πολιτών ε, ε, αν θέλουν να παντρευτούν ή ίσως για κάποιον άλλο λόγο να μετικήσουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος να μπορούν να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Είναι ένα ουσιαστικό πρόβλημα των πολιτών και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν βέβαια και αμφισβητήσεις. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, χρειάζεται χρόνο, υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και και παραδόσεις και θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη αναγνώριση των επαγγελμάτων και γι' αυτό δεν ε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε όλα τα επαγγέλματα ε, κατευθείαν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά θα πρέπει επίσης να ερευνήσουμε τι γίνεται και πιστεύω ότι εδώ βοηθάει και το Solvit. Δηλαδή αν υπάρχουν λάθος στις δομές στο σύστημα και πώς μπορούμε να υπάρξουν βελτιώσεις. Το θέμα δεν θα κλείσει ποτέ. Είναι ένα πρόβλημα διαρκείας, διότι υπάρχουν συνεχώς νέα επαγγέλματα, νέα, ε, επαγγελματική, κατάρτιση και γι' αυτό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη χρειάζεται, χρειάζεται καλή θέληση και κάνω έκκληση γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λέχνερ. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι η κυρία Γκέπχαρτ. Για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να παρατηρήσω ότι είναι απίστευτη εσχήνη το ότι δεν έχουμε επίτροπο άντρα ή γυναίκα εδώ παρόντα ή παρούσα. Διότι εδώ πρόκειται για ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προσβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απαράδεκτη υπόθεση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Ναι, δεν σηκώθηκε όμως. Λυπούμε, δεν τον είδα. Εντάξει. Τι να πω. Έστω, δεν μπορώ να δεχτώ μια τέτοια κατάσταση. Αλλά για να περάσω στο θέμα αυτό, στο θέμα το οποίο μας απασχολεί πράγματι. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές συνάδελφοι, Πρόκειται για τους, την ηθαγένεια, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ασκούν το επάγγελμά τους εκεί όπου ζουν, εκεί όπου διαμένουν και εκεί όπου πραγματικά θέλουν να εργαστούν. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την νομοθεσία, αυτούς τους νόμους, για να διευκολύνονται οι πολίτες και μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους να μπορούν να εργάζονται με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό είναι ανήκουστο πράγματι ότι κράτη-μέλη σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν αναλάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε αυτή η νομοθεσία να εκτελεστεί, να εφαρμοστεί και να μεριμνήσουν έτσι ώστε η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών θα μπορεί να διασφαλίζεται. Και πρέπει λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδιαίτερη προσοχή και με ιδιαίτερη μέρημνα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμα. Ένα σημείο θέλω να υπογραμμίσω που είναι σημαντικό και που ως Κοινοβούλιο το έχουμε αναφέρει επανειλημμένα. Πρέπει να μεριμνήσουμε ότι τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά επαγγελμάτων πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να έχουν κάτι στα χέρια τους οι Ευρωπαίοι πολίτες και να μπορούν να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν οργανώσεις που μεριμνούν γι' αυτό αλλά θα ήταν κάτι το σημαντικό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το θέμα ώστε αυτό να προαχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον Κριστιαν Μπουζόη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό συμπεριλαμβάνει την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών που είναι θεμελιώδου σημασία για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όπως είπαν οι συνάδελφοι πιο πριν, παρόλη την οδηγία που υιοθετήθηκε το 2005 επαγγελματίες που θέλουν ελεύθερα να κυκλοφορήσουν να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προσκόμματα. Είδα πολλές τέτοιες περιπτώσεις προσωπικά που μου ε, πέσαν την προσοχή μου ε, πολίτες από τη Ρουμανία όσον αφορά και τα πιο διαφορετικά επαγγέλματα. Ήμουν και εισηγητής ε, όσον αφορά το δίκτυο Solvit και όπως προαναφέρθηκε ήδη ένα μεγάλο τμήμα των περιπτώσεων που πρέπει να επιλύει το Solvit συσχετίζονται με δυσλειτουργίες στο σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών πιστοποιητικών και ε, ικανοτήτων και πρέπει να δούμε αυτό σε βάθος, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Είναι θεμελιώδες να έχουμε καλύτερη επικοινωνία και επαφές ε, μεταξύ των συνδέσμων για να έχουμε προσέγγιση των κρατών μελών και κατανόηση, να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη πώς λειτουργούν τα άλλα συστήματα, να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας για να αντιμετωπιστούν και να αρθούν ε, προσκόμματα και εμπόδια επιθυμούμε τα πέντε κράτη τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τις τελικές διατάξεις της οδηγίας ή κράτη-μέλη που δεν έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά την οδηγία να μπορέσουν να δικτυωθούν καλύτερα ώστε να επανορθωθεί αυτή η κατάσταση πραγμάτων. Οι υπηρεσίες λοιπόν πρέπει να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών ικανοτήτων. Ευχαριστώ κυρία Ρούιλε, παρακαλώ δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό το στόχο. Όλοι θέλουμε φυσικά οι πολίτες, γυναίκες και άνδρες να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ένωση και να μπορούν να ασκούν τα επαγγέλματά τους ελεύθερα. Το ζήτημα είναι φυσικά γιατί αυτή η οδηγία μετά από τέσσερα χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί σωστά σε λίγο θα είναι πέντε χρόνια και νομίζω έχει νόημα ως Επιτροπή όχι μόνο στην προπαρασκευή των, ε, της νομοθεσίας να συνεργαζόμαστε αλλά να κάνουμε και ανάλυση στη συνέχεια ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις. Η αναγνώριση επαγγελματικών πιστοποιητικών και ικανοτήτων δεν είναι η μόνη οδηγία που δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό είναι ένα, ένας κόδωνας κινδύνου που ακούμε ότι εδώ σημαίνει και δίνει ένα μήνυμα. Να δούμε Ποια είναι τα προβλήματα, σε τι οφείλεται αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν διαφορετικά αίτια. Αφενός, για να το πούμε απλά, τα κράτη-μέλη διστάζουν. Έχουν κάποιες προστατευτικές τάσεις. Υπάρχουν τέτοιοι λόγοι. Όμως υπάρχουν και εξειδικευμένοι λόγοι διαφορετικών παραδόσεων, διαφορετικού πολιτισμού και νομικών συστημάτων και διαφορετικής νομολογίας. Και σε αυτό πρέπει πάλι να επικεντρωθούμε. Πρέπει να δούμε αν η οδηγία ακριβώς ε, πετυχαίνει αυτό που θέλαμε να πετύχει ή αν κάποια πράγματα δεν μπορούν να επιτευχθούν από πλευρά τη. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Η εξ άντε, η εκ ανάλυση είναι ένα από τα σημαντικά θέματα στη συζήτηση αυτή που θα γίνει, που πρέπει να απασχοληθεί η Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή και να δώσει συνέχεια σε αυτά. Έχουμε ερωτήσει και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με εκπλήσει γιατί αυτό ο οδηγό τώρα δημοσιεύεται μετά από τέσσερα χρόνια. Αυτό το εγχειρίδιο ή ο οδηγό θα έπρεπε πριν από χρόνια να έχει δημοσιευθεί. Το χαιρετίζω, είναι επικοδομητικό το ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε. Όμω πριν από χρόνια έπρεπε να είχε γίνει γίνει αυτό. Προσθέτω τη φωνή μου στην ε, ερώτηση της κυρίας ε, Γκέπχαρντ. Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά πιστοποιητικά. Αυτό είναι το αναγκαίο δεύτερο βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα για ένα μισή λεπτό στον κύριο Μπίλαν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε περίοδους κρίσης, σε περίοδους που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τώρα, είναι πολύ σημαντική η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς. Δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή την ενιαία εσωτερική αγορά. Δεν θα ολοκληρωθεί χωρίς την ελευθερία κυκλοφορίας, που διασφαλίζεται μεταξύ άλλων και από αυτή την οδηγία. Γι' αυτό είναι ανησυχητικό ότι μετά από τέσσερα χρόνια, μετά από έγκριση αυτής της οδηγίας, εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται στα κρατη Και αρκετά σε σχέση με, την ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2007 που προβλεπόταν από την οδηγία δεν τήρησαν. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είσαστε υπερβολικά παθητικοί και αδρανοί στα τελευταία χρόνια. Τι κάνατε σε σχέση με τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν έγκαιρα να υλοποιήσουν αυτή την οδηγία. Δεύτερο πότε θα δημοσιεύσετε μια έκθεση με την αποτίμηση των πραγμάτων για την εφαρμογή, την εκτέλεση αυτής της οδηγίας και ποια θα είναι η βάση για συμπεράσματα τα οποία θα συναρθούν από κοινού σε σχέση με την έκθεση. Κατά τέλη του έτους η οδηγία περιπηρεσιών θα πρέπει να υλοποιηθεί. Ξέρουμε ότι πολλά κρατημέλη δεν θα τα καταφέρουν να έχουν έγκαιρα την νομοθεσία έτοιμη ώστε να γίνει αυτό. Ποια, ποια συνάρτηση βλέπετε μεταξύ των δύο οδηγιών και όσον αφορά και την ε, κινητικότητα των ε, νοσηλευτριών, των νοσοκόμων για την Πολωνία, σημαντικό θέμα. Και σε σχέση επίσης και με την εισαγωγή διατάξεων για την κατάρτιση των ε, νοσηλευτριών, των νοσοκόμων. Θα ήθελα να μου πείτε ποιε διατάξεις, ποια διαβήματα κάνατε ώστε να υποστηριχθούν οι νοσοκόμοι από την Ανατολική Ευρώπη και από την Πολωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στον Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα ευχαριστώ που μα δίνετε την ευκαιρία να εκφράσουμε την απόψη μα. Θέλω να πω ότι μετά από τη διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπής και Κοινοβουλίου και τότε με την οδηγία περί που πριν ε, από μήνε είχαμε συζητήσει εκτενώς, το είχα δει, ότι ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχει ο αρμόδιος επίτροπος που θα επιλαμβάνεται αυτού του θέματος. Νομίζω ότι τώρα με την Επιτροπή δεν έγινε αυτό, αλλά θέλω να απευθύνω έκκληση προς την Επιτροπή και στους εκπροσώπους της. Αυτό το τμήμα της Διοργανικής Συμφωνίας το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και γιατί, όχι μόνο για τυπικούς λόγους, διότι επειδή για αυτό το θέμα πρόκειται για μια κέρια πολιτική υπόθεση θεμελιώδου σημασία για του πολίτες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα οικονομικά θέματα, οικονομικά πολιτικά θέματα, ο συνάδελφο ανέφερε την οδηγία περί υπηρεσιών, μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν υπάρχουν αμοιβέ αναγνωρίσει επαγγελματικών ε, σπουδών και πιστοποιητικών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως πολλοί άνθρωποι αμήχανα αντιμετωπίζουν την κατάσταση όταν βλέπουν ότι μεταξύ εργοδοτών δεν υπάρχει μια ενιαία κατάσταση αντιμετώπισης των εργαζομένων όσον αφορά τα πιστοποιητικά αυτά και την αναγνώρισή τους. Αυτοί οι άνθρωποι σε μια ολόκληρη σειρά σε μεθοριακές περιοχές, περιοχές μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας για παράδειγμα αλλά αυτή δεν είναι η μόνη προβληματική περιοχή μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ανήμποροι τελείως αμήχανοι και κανείς δεν τους βοηθάει πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες όταν τέτοια προβλήματα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και στο μέλλον θα πρέπει λοιπόν εδώ και το ανέφερε ο εισηγητής μας Κουρτ Λέχνερ να λάβουμε υπόψη αυτά τα πράγματα είναι έργο μας αυτούς τους πολίτες να τους πάρουμε στα σοβαρά στα αιτήματά τους. Και σε αυτό ανήκει πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει την αναγκαία σημασία σε αυτό το ζήτημα. Ελπίζω ότι με τη νέα Επιτροπή θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να προαγάγουμε αυτό το ζήτημα. Και παρακαλώ στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής να διαβιβάσετε αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Μπερναντέτ Μπενιό για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ήδη έχουμε συζητήσει για τους ε, φόβους που έχει δημιουργήσει η οδηγία των υπηρεσιών και εδώ βλέπουμε ε, για την ε, οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελμάτων ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη σε εθνικό επίπεδο και αν βασίζεται εκεί η αμοιβαία αναγνώριση δεν αναγνωρίζονται ορισμένα επαγγέλματα. Να αναγνωρίζονται λοιπόν Λοιπόν, τα ε, επαγγέλματα χωρίς να υπάρχει ε, μία ενιαία αντιμετώπιση και προσαρμογή της ανωτάτης παιδείας δεν μπορεί ε, να βοηθήσει τους πολίτες και το πιο βασικό αναφέρεται σε τα προβλήματα των ιατρικών επαγγελμάτων και αναφέρουμε εδώ στη χώρα μου που ίσως δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα σε άλλες χώρες η ΑΜΕΑ χρειάζεται ειδική ε, ε, ε, επιμόρφωση για να μπορέσει να δουλέψει στη Γαλλία. Πρέπει λοιπόν να βασιζόμαστε στην ευρωπαϊκή ιδέα αλλά να συμπληρώσουμε τις διατάξεις για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα επαγγέλματα για τα οποία οι γλωσσικές γνώσεις και η εναρμόνιση των γνώσεων επιβάλλεται. Υπάρχει μια θαυμάσια πρωτοβουλία από όλου τους υπευθύνους υγείας για μια ευρωπαϊκή κάρτα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους υπευθύνους και θα έπρεπε να επεκταθεί η χρήση της για να μπορέσει να προκαλέσει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο για ένα λεπτό και μισό στην κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν συζητάμε την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την καλή λειτουργία τη εσωτερική αγορά, πρέπει να δούμε τη τρέχουσα κατάσταση στον ε, ε, τομέα της, ε, στο τομίσο που πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Επιπλέον, αυτέ τι οδηγίε πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω μέτρα για την αμοιβαία αναγνώριση όχι μόνο των διπλωμάτων, αλλά και όλων των άλλων επαγγελματικών ε, ε, προσόντων στον τομέα της υγείας. Απαιτούνται γλωσσικά προσόντα, αλλά περισσότερο από όλα χρειάζεται υψηλό επίπεδου ε, φροντίδα. Νομίζω, νομίζω ότι απαιτείται μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα επαγγέλματα της υγείας μέσω μιας κοινή βάσης δεδομένων, παραδείγματος χάρη. θα πρέπει να σκεφτούμε κοινά πρότυπα για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η κινητικότητα των επαγγελμάτων υγείας είναι θέμα και δημόσιας υγείας. Ε, θα πρέπει να ε, έχουν ήδη εφαρμοστεί, ε, υιοθετηθεί επιπλέον κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εμπορευμάτων. θα πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο για, την, για τις υπηρεσίες της υγείας. Όταν οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν αφιλεγόμενε πρακτικές όπως είναι η ηλεκτρονική ε, παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαίω την κινητικότητα των επαγγελμάτων τη υγεία, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε πρόσβαση στι υπηρεσίε υγεία, έγκαιρε υπηρεσίε υψηλή ε, ποιότητα. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλου μα και ελπίζω ότι και τα κρατημέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν ε, σοβαρά το γεγονό ότι κάποια συστήματα υγεία έχουν ε, μείνει χωρί επαγγελματίε και δυσκολεύονται πάρα πολύ να δώσουν και τι βασικέ διαφορετικές ακόμα υπηρεσίες υγείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει για δύο λεπτά η κυρία Χάντσλικ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε να έχουν κινητικότητα οι πολίτες μας, Πρέπει να είναι σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή αποκτήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα στην Πολωνία, παραδείγματο χάρη, ότι δεν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εμπόδια σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μέλος. Και ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει μια πληθώρα διαφορετικών ε, κανονισμών για όλα αυτά τα επαγγέλματα. Αυτή είναι μια πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους πολίτες. Η πρόκληση όμως πραγματική είναι να βρουν τον δρόμο τους μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο αυτού του πολύπλοκου συστήματος. Ε, αυτή η οδηγία λοιπόν είναι μόνο μία διάσταση της όλης συζήτηση. Ας μην ξεχνάμε ότι προβλήματα δημιουργούνται επίσης και λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης ε, ε, των κρατών μελών για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων κρατών μελών. Επίσης, η ε, διοίκηση, η εθνική διοίκηση πρέπει να ευλακεί περισσότερο την τελευταία φορά συζητήσαμε το, την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα η οδηγία αυτή θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα και όχι να είναι ακόμα ένα εμπόδιο για την ε, ε, κοινή αγορά, για την εσωτερική αγορά. Κυρίες και κύριοι, σε δέκα μέρες περίπου ε, η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτές οι δύο οδηγίες είναι συμπληρωματικές από κάποιες απόψεις. Η εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα δεν είναι ε, και πολύ επιτυχημένοι. Σας παρακαλώ λοιπόν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και οι δύο αυτές οδηγίες γιατί τις χρειαζόμαστε για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κορέιεντε Ντεκάμπος για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αν η αναγνώριση των επαγγελματικών πιστοποιητικών σε μία ενιαία νομοθετική πράξη παγιώθηκε και εκεί 15 οδηγίες συμπτύχθηκαν πράγμα το οποίο ε, δημιουργήσε προβλήματα στην εφαρμογή όσον αφορά τα διάφορα κρατημέλη. Είναι γνωστές οι δυσκολίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να σημειώσει τα σημεία αυτά και να κάνει μία ανάλυση των προβληματικών πεδίων που υπάρχουν στην εφαρμογή αυτού του πολύ σημαντικού ε, πεδίου διάταξη για την ενιαία εσωτερική αγορά η προστατευτική τάση που παρουσιάζεται σε διάφορα επίπεδα αποτελεί ένα εμπόδιο όχι μόνο για την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αλλά και για την ενιαία εσωτερική αγορά. Πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν, ε, τα θέματα που δημιουργούν προβλήματα ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση αυτών θα πρέπει από πλευρά του να κάνουν τη δουλειά του τα κράτη-μέλη. Αλλά πρέπει να γίνει και η προσπάθεια να διευκολύνουμε αυτή την τάση όσον αφορά τις επαγγελμα... τα επαγγελματικά πιστοποιητικά. Η βελτίωση αυτή τη οδηγία θα πρέπει να περάσει από την δια... ανακοίνωση και διάχυση των διαδικασιών και όσον αφορά το δίκτυο αυτό για την αναγνώριση των πιστοποιητικών και την εφαρμογή και την λειτουργία συνδετικών σημείων, συνδέσμων για να μπορέσει να υπάρξει η σωστή εφαρμογή αυτής τη οδηγία όσον αφορά και την οδηγία περιπηρεσιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. επόμενο είναι ο κύριος Γκρέχ για ένα λεπτό. Κύριε, Κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ε, εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μία έλλειψη ενδιαφέροντος στα κράτη-μέλη και αυτό οφείλεται εις τον ε, αντιμαχόμενο τρόπο με τον οποίο ε, αντιλαμβάνονται την εσωτερική αγορά τα διάφορα κράτη διότι λέγεται ότι σέβονται την κοινή αγορά αλλά όχι μία συνεπή εφαρμογή ε, πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζουν τα κράτη και πώς εφαρμόζουν αυτή την οδηγία να έχουμε ένα σημείο αναφοράς για όλα τα κράτη-μέλη οπότε το κάθε κράτος μέλος να μπορέσει να προσθέτει τις πληροφορίες κατά τρόπον ώστε η οδηγία αυτή να μπορέσει ε, πραγματικά να ε, εφαρμοστεί. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρόγραμμα έχει για την εφαρμογή αυτή της οδηγίας και αν επιθυμούν να προωθήσουν την ιδέα της ενιαίας αγοράς και να μην το αντιμετωπίζουν όπως όλοι. Η κυρία Κάτριν Στίλερ είναι η επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σήμερα το πρωί μιλήσαμε πολύ για το Solvit και στην τελευταία επιτροπή ΙΜΚΟ μιλήσαμε και για τη χρηματοδότηση των κέντρων Solvit και ο κύριος Μπανιέ θα έπρεπε ίσως να το σημειώσει πριν ε, την ακρόασή του αλλά ε, θα πρέπει το Solvit να μπορεί να συνεχίσει να μας προσφέρει τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρει και τώρα. Υπάρχουν ε, διάφορα επαγγέλματα που κινδυνεύουν, ιδίω τα επαγγέλματα σε σχέση με την υγεία που μπορούν να προκαλέσουν θανάτους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία σωστή ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με ε, τις ε, διατάξεις κατά τρόπον ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία. Χρειάζεται μία ανταλλαγή πληροφοριών αλλά θα πρέπει κάποιος να είναι εγγεγραμμένος σαν υποψήφιος για να τεθεί το ερώτημα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ενιαίος τρόπος καταγραφής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις προτάσεις που κάνατε. Ευχαριστώ και τώρα θα προχωρήσουμε στην διασία catch the eye, δηλαδή ε, ε, αυθόρμητες παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Μέχρι στιγμής έχουμε έξι υποψηφίους εγγεγραμμένους και αν ε, όλοι σεβαστούν το χρόνο θα μπορέσουν να μιλήσουν. Πρώτο ο κύριος Φιλίπ Μπενζουρίν. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, πολλά έχουν λεχθεί για την αμοιβαία αναγνώριση των των επαγγελματικών ε, ικανοτήτων και το θέμα είναι ε, γιατί κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν τόσο δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί και αυτό οφείλεται στην περιπλοκή της στην καθημερινή εφαρμογή. Υπάρχουν τρεις δυσκολίες. Πρώτον τις γλώσσες που αναφέρθηκε. Δεύτερον η περίπλοκη διαδικασία για την αναγνώριση του εγκύρου ενός διπλώματος χρειάζεται δηλαδή ε, μεγάλη προσπάθεια για να αναγνωριστεί το αρχικό δίπλωμα και υπάρχει ετερογένεια των αρχικών καταρτήσεων και επ' αυτού θα θεωρούσα ότι θα ήταν καλό η Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη-μέλη για κάθε επάγγελμα ε, να ζητήσει ε, να υπάρχει μία ενιαία αρχή η οποία θα αναλάβει την ε, συνεχή κατάρτιση για να μπορούν οι υπεύθυνε αρχές να ε, συγκεντρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καταρτήσουν ένα κοινό πίνακα ε, γνώσεων κατά τρόπον ώστε να υπάρχει μία ενιαία συνεχής επιμόρφωση. Ευχαριστώ. Ο Μάρκ Ταραμπέλα για ένα λεπτό. <coughs> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Βέλγιο είναι ένα από τα πέντε κράτη-μέλη που δεν έχουν μεταφέρει ακόμα αυτή την οδηγία. Αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, δεν του μένει παρά να λύσει το πρόβλημα των επαγγελμάτων του ταξιδιού. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα γενές στο βελικό σύστημα όσον αφορά την μεταφορά ε, του, των οδηγιών, αλλά φαίνεται ότι και η οδηγία αυτή συγκεκριμένη είναι ιδιαίτερα ε, περίπλοκη. Μία κακή ή μερική ε, εφαρμογή πάντως και μεταφορά δεν είναι ένα πρόβλημα που περιορίζεται μόνο στο Βέλγιο. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση στην Κομισιόν να λύσει αυτό το πρόβλημα για την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών που είναι ο βασικός στόχος αυτής της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαμέσκη για την καλή του δουλειά. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα δεν ε, ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ευρύτερα. Ε, αυτό ζητούσαμε πρόσφατα με την καναδική αντιπροσωπεία, ότι είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πρέπει όμω να είμαστε ουτοπιστέ. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η τα επαγγελματικά προσόντα ε, θα ε, βρίσκονται, θα τη χάνουν μεταχείρισης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν ιστορίες που ε, μας λένε ότι όταν δεν έχουν ε, την ικανότητα να περάσουν ένα μάθημα κάποιοι φοιτητέ, πηγαίνουν σε ένα άλλο κράτο μέλο και περνάνε εκεί αυτό το μάθημα. Πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχουν στάνταρ που να είναι τα ίδια παντού. Γιατί ε, διαφορετικά δεν θα επιτύχουμε το επιθυμητό επίπεδο ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών και, και τη εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κέλλη. Δίνω το λόγο σε έναν άλλον κύριο Κέλλη, τον άλλον Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην σας μπερδεύουν αυτοί οι δύο Κέλλη πάρα πολύ. <clears throat> Όσον αφορά την ε, ε, ε, μη μεταφορά της οδηγίας αυτής στα κράτη-μέλη, αυτό μας κοστίζει θέσεις εργασίας. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Το διασυνορικό εμπόριο στην εσωτερική αγορά δεν είναι καθόλου αυτό που θα έπρεπε να είναι πρέπει να ενισχύσουμε το διασυνολικό ε, εμπόριο και πρέπει να περάσουμε σε νέους τομείς επιχειρηματικότητας ε, για να προωθήσουμε τα πιο πρωτοπόρα προϊόντα. Η εξαγωγή υπηρεσιών σε χώρες όπως η Ιρλανδία είναι ένας νέος ε, πολλά υποσχόμενος τομέας. Μέχρι τώρα η μη συμφωνία των κρατών μελών να συμφωνήσουν για αυτού του κανόνε περιορίζει την ικανότητά μα να πουλήσουμε τι υπηρεσίε μα ε, σε διασυνοριακό επίπεδο. Και αυτό ε, περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη δεν, δίνουν, ε, δεν δείχνουν αρκετό σεβασμό για τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται. Πρέπει η Κομισιόν να εντοπίσει τα εμπόδια που εμποδίζουν την ε, <clears throat> υλοποίηση της ε, ε, νέας αγοράς για τους λόγους αυτούς. Φανίστε Ρόι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο μία πτυχή σε αυτή τη συζήτηση αυτών των θεμάτων θα ήθελα να υπογραμμίσω. Περί τι πρόκειται εδώ. Εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες απουσιάζουν εν μέρη εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά ένα εμπόριο πιστοποιητικό πιστοποίησης ε, ικανοτήτων ξεκινά. Μπορούν να υπάρξουν κίνδυνοι που ελοχεύουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία. Παράδειγμα, στον τομέα της ασφάλειας, ε, αν μια μεγάλη επιχείρηση όπως κάποια χημιοβιομηχανία ή άλλη μεγάλη επιχείρηση, τι συμβαίνει. Οι εθνικές εποπτικές αρχές για κάποιες κατηγορίες ε, δεν επαρκούν. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο, το γνωρίζετε ότι συμβαίνει αυτό ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την περίπτωση και τι μπορεί να αλλάξει. Γιατί είναι πολύ προβληματικό. Είναι ένα επιθύμητο φαινόμενο αυτό το οποίο πρέπει να πάψει να υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τσφέρ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αντιμετωπίζουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών και επαγγελματικών διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα, διότι τα πιστοποιητικά προέρχονται από τα <clears throat> εκπαιδευτικά συστήματα και είναι 27 διαφορετικά συστήματα αυτά μέσα στα κράτη-μέλη. Ε, και θα θυμόσαστε ότι τον Μάρτιο εγκρίναμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει ώστε τα, ε, τα συστήματα παιδείας και εκπαίδευσης να μπορούν να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Όμως αυτό το πλαίσιο έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να το εκτελέσουν, να το εφαρμόσουν σωστά. Κάποια το εφάρμοσαν εν μέρη. Κάποια άλλοι απλά και μόνο για να προσπαθήσουν να μεταθέσουν κάποιες ε, διατάξεις. Όμως, περιπτώσει στο μέλλον όσον αφορά τα κράτη-μέλη πολύ μεγάλο έργο απομένει να επιτελεστεί και να καλυφθεί για αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο πιστοποιητικό και επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πρώτον, πρέπει να εφαρμοστεί σωστά αυτό το πλαίσιο, γιατί με την αναγνώριση θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ε, τώρα, για να τελειώσουμε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαμέσκη εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε ε, προς εσάς και ε, προς τους ευρωβουλευτές που δεν σηκώθηκα την πρώτη φορά αλλά ε, δεν έχω αρκετή πείρα και ήταν και νωρίς το πρωί. Καταρχήν θα ήθελα λοιπόν να απαντήσω σε ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηρίξει τα κράτη-μέλη για να ετοιμάσουν την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της οδηγίας και όταν τελείωσε η έχουμε πίεση ε, ε, για την εφαρμογή ε, βοηθήσαμε με έναν οδηγό και υπάρχουν τώρα οδηγίες προς όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε έναν κώδικα συμπεριφοράς για, τις, για διοικητική συμπεριφορά που κυκλοφόρησε φέτος Πέρυσι τα ε, ε, κράτη που δεν είχαν συμμορφωθεί προσήχθησαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχουν τώρα έξι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την έλλειψη ε, εφαρμογής της οδηγίας σε κράτη-μέλη και έχει ξεκινήσει διαδικασία κυρώσεων και υπάρχει συγχρόνως όμως και ένας οδηγός για τους επαγγελματίες επί των διατάξεων. Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω όλους όλους και ιδίως τον πρόεδρο της Επιτροπής Μάλκολμ Χάλμορ για τη σημαντική του συνδρομή και πιστεύουμε ότι τώρα το μπαλάκι είναι στα κράτη-μέλη. Αυτοί θα πρέπει να ε, προσαρμοστούν και να μπορέσουν ε, να το πράξουν υπό την παρακολούθηση του Κοινοβουλίου για να γνωρίζουμε πώς εφαρμόζεται η οδηγία και πώς είναι δυνατόν να επηρεάσει την εξέλιξη του επαγγελματικού περιβάλλοντος στα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και κατά αυτόν τον τρόπο φτάσαμε στο τέλος της συζητήσεώς μας και τώρα επιτρέψτε μου σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη να περάσουμε στο δεύτερο θέμα ε, για την πολιτική συνοχή μετά το 2013. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στη συντάκτρια την κυρία Ντανούτα Μαρία Χιούμπνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πίτροπη.